Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίσω την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης. Πρώτο σημείο της μερίσιας διάταξης είναι οι ψηφοφορίε επί των αιτήσεων Να Με το άρθρο 154 του κανονισμού έχουμε τρεις ε, αιτήσει. Η πρώτη από την Επιτροπή Αλία σε σχέση με τους κανόνες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση. Μπορεί να ε, μιλήσει ένας ε, υπέρ της ε, πρότασης ή ο πρόεδρος Επιτροπής, η συγητής, και δύο. Ποιος θα ήθελε το λόγο? Κανείς από ό,τι φαίνεται ούτε κατά. Θέλει κάποιο να ψηφί, μιλήσει, οπότε ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αύριο από τις 12 και μετά θα γίνει η ψηφοφορία 12 ε, μάλλον ε, στις ε, μία το μεσημέρι λίγη προθεσμή για την κατάθεση τροπολογιών σήμερα. Και τώρα έχουμε το δεύτερο θέμα, άδειες αλίας για ληφτικά σκάφη της Ένωσης, ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου και αληφτικές δραστηριότητες αληφτικών σκαφών του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα της Ένωσης. οι δυο. Ποιος θα ήθελε το λόγο, αν κάποιος θέλει το λόγο. Πριν ψηφίσουμε, ουδής. Επομένως, μπορούμε να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, εποχές εγκρίνεται και για αυτό το αίτημα αύριο από τις 12 και μετά θα γίνει ψηφοφορία και για την κατάθεση τροπολογιών σήμερα στη μία λίγη προθεσμία. Τρίτο αίτημα από την Επιτροπή Μεταφορών για ορισμένε πτυχέ ασφάλεια των σιδηροδρόμων και τη συνδεσιμότητα όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασίλειου τη Μεγάλη Βρετανία και τη Βόρεια Ιρλανδία από την Ένωση. ίδιο, ίδια διαδικασία. Θα ήθελε κάποιο το λόγο, Όχι. Όχι. Δεν θέλει κάποιο το λόγο. Ωραία. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Και αυτό το αίτημα γίνεται δεκτό. Δεν το εννοείται αυτό φαντάζομαι. Λοιπόν, αύριο από τις 12 θα ξεκινήσουν ψηφοφορίες και θα ψηφιστεί και αυτό το θέμα και μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες μέχρι σήμερα στη μία το μεσημέρι. Επίσης θα ήθελα να σας πω ότι συμφώνησαν οι πολιτικές ομάδες σε ό,τι αφορά το ψήφισμα που θα ολοκληρώσει τη συζήτηση για τη δήλωση της Αντιπρόεδρου Κομισιόν και είπα της εκπροσώπου ε, ε, σε σχέση με την κατάσταση εκτάκτης ανάγκης ε, στη Βενεζουέλα. Το ψήφισμα λοιπόν να μην ψηφιστεί σε αυτήν αλλά στην επόμενη σύνοδο Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, φαντάζομαι γίνεται δεκτό αυτό. Επόμενο σημείο Έχουμε δήλωση ε, για την ισορροπία των φύλων κατά το διορισμό σε ενωσιακέ θέσει του οικονομικού και νομισματικού τομέα. Δηλώσει τη Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξ ονόματο του Συμβουλίου, η κυρία Τσιότ, έχει πρώτη το λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όσοι δεν θέλετε να ακούσετε την παρέμβαση αυτή, να αποχωρήσετε γρήγορα από την αίθουσα. Κύριε Φερχόφστατ, κύριε Μπούλμαν, εδώ δεν έχουμε πηγαδάκια. Κύριε Σφάπ, παρακαλώ. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους Τι γίνεται από την πλευρά των πέντε αστέρων, έχουν φτιάξει εδώ ένα τείχο στην αίθουσα. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε Τσιώτα, έχετε τώρα το λόγο. Καλημέρα. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ταγιάννη για την επιστολή του που έλαβε το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Να σας διαβεβαιώσω ότι δεσμευόμαστε να προαγάγουμε την ισορροπία των φύλων. Πρόκειται για σημαντικό θέμα. Η ισορροπία των φύλων και η τοποθέτηση γυναικών σε υψηλέ θέσει είναι προτεραιότητα. Όλα αυτά βασίζονται σε κανόνε που οφείλουμε να σεβαστούμε. Το Συμβούλιο ανέκαθεν έδρασε και θα συνεχίσει να δρά βάσει των σχετικών διατάξεων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, της Ενωσιακής Νομοθεσίας όσον αφορά τους διορισμούς. Εκτιμώ ότι και όλα τα άλλα όργανα θα δράσουν εντός του νομικού πλαισίου και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να προαγάγουν την ισορροπία των φύλων. Βάσει όλων αυτών εκπλήττωμε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει ξανά το θέμα έναντι του Συμβουλίου. Η επιστολή Ταγιάννη αναφέρεται σε νομικές πράξεις που ρυθμίζουν τις τοποθετήσεις στα τρία όργανα της Ένωσης και συγκεκριμένα το ενιαίο συμβούλιο, η τραπεζική αρχή και η ενιαία αρχή για τις τράπεζες. Το Συμβούλιο δεν εμπλέκεται στην κατάρτιση του καταλόγου των προσδιορισμό ατόμων. Ο τελικός κατάλογος για τους διορισμούς στο Συμβούλιο ρύθμιση των ε, τραπεζών είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και για τα δύο αυτά συμβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφασίζει επί των επιτυχόντων. Ο ρόλος του Συμβουλίου λοιπόν περιορίζεται στην τυπική έγκριση των ε, διορισμών, των τοποθετήσεων του Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, το Συμβούλιο δεν έχει κανέναν ρόλο να διαδραματίσει όσον αφορά την επιλογή τώρα των μελών τη Εκτελεστική Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Συμβούλιο όντω διαδραματίζει ρόλο στην διαδικασία επιλογή. Να σα διαβεβαιώσω ότι εμεί συνεχίζουμε να υπογραμμίζουμε την σημασία τη ισορροπία των φύλων σε κάθε διαδικασία επιλογή και καλούμε τα κράτη-μέλη να προτείνουν γυναίκε ω υποψηφίου θεωρώ βέβαιο ότι όλα τα ενωσιακά όργανα τα οποία εμπλέκονται στην κατάρτιση των καταλόγων υποψηφίων σέβονται την αρχή της ισορροπίας των φύλων και ότι θα συνεχίσουν να το πράττουν στο μέλλον. Ως Προεδρία του Συμβουλίου η Ρουμανία θα συνεχίσει να προάγει σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αρχή της ισορροπίας των φύλων για να διευκολύνει τον διάλογο για τις μελλοντικέ διαδικασίες. Για να προαγάγουμε λοιπόν την μας, νομοθετικό μας θεματολόγιο βάσει της σχετικής οδηγίας για την ισορροπία των φύλων. Στον τομέα αυτόν έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος χάρη στι συνεπείς προσπάθειες και του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει και τις οδηγίες για την ισορροπία εργασιακής ζωής και οικογενικής ζωής. Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προωθήσουμε το θέμα της ισορροπίας των φύλων για να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον ισόρροπο στην εσωτερική μας αγορά μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσιώτεκ. Μέρος τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Γιούροβα. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι βουλευτέ, εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των οποίων και ο κύριο Αντιπρόεδρο Ντομπρόφσκη και Μοσκοβισή, στι Βρυξέλλε σήμερα στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ε, θα έχουν την ευκαιρία και εκείνοι να συζητήσουν το θέμα αυτό και θέλω και εγώ να σα ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή. Ο πρόεδρο Γιούνκερ απήντησε χθε στην επιστολή του πρόεδρου Ταγιάννη για το θέμα αυτό. Κατά πρώτον, να υπογραμμίσω ότι αυτή η Επιτροπή ε, είναι ταγμένη στο σκοπό της ισότητας των φύλων και έχει αναλάβει αποφασιστική δράση προς το σκοπό αυτό. 69,6% μάλλον 39,6% των, ε, των στελεχών των επιχειρήσεων είναι γυναίκες, από 30% το 2014. Φτάσαμε από το 14% στο 30%. Και από το 5% στο 12%. Ο αριθμός των γυναικών, των γυναικών διευθυντριών έχει φτάσει στο 42%. Ενώ είχαμε μια αναλογία 3 προς 20. Επίσης, ε, διοικητικέ θέσεις στον τομέα των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, οι γυναίκες εκπροσωπούν μόνο το 15% των στελεχών η υποεκπροσώπηση των γυναικών έχει παρατηρηθεί και στον δημόσιο τομέα. Όσο νωρίτερα δράσουμε, τότε θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι για τους φορείς των ε, κεντρικών τραπεζών των εθνικών κρατών. Αυτή η χαμηλή εκπροσώπηση έχει επίσης ε, την ε, ίδια συχνότητα και στα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμούς. Η που υποψήφοι είναι τετραπλάσια από ότι γυναίκε Για τι συγκεκριμένε υποθέσει που σήμερα μα απασχολούν, να πω ότι ότι από το άρθρο 283 κάθετος δύο της ε, συνθήκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανέναν ενεργό ρόλο να αναλάβει στον διορισμό των ε, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας. Ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, ο ρόλος της, Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιορίζεται στο να συνδράμει τον, ε, ε, το Σύνολο Συμβούλων στην επιλογή και το διορισμό του Προέδρου και του Προεδρείου στον μηχανισμό εξυγίανσης που αυτή τη στιγμή πρόεδρος είναι γυναίκα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς μπορεί να δώσει ένα κατάλογο υποψηφίων ε, στο Κοινοβούλιο για τι θέσει των Προέδρων, Αντιπροέδρων και των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να επιλέξουν. Βάσει του σχετικού κανονισμού για τον ορισμό του Συμβουλίου, θα πρέπει οι δεξιότητες, οι γνώσεις και τα προσόντα των υποψηφίων, καθώς και η εμπειρογνωμοσύνη του να είναι το κριτήριο για την επιλογή του. Επίσης, Βάσει του άρθρου 56.4 του κανονισμού, οι υποψήφοι πρέπει να επιλέγονται βάσει ενός ανοιχτού ε, μια ανοιχτή διαδικασία επιλογή που να σέβεται τι αρχέ τη ισότητα των φύλων, τη πείρα και των επαγγελματικών προσόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ τη υποστήριξη των γυναικών για τι σχετικέ ε, θέσει. Θα πρέπει να Σεβαστούμε όμω και το νομικό πλαίσιο των διαδικασιών επιλογή. Γι' αυτό έχουμε τηρήσει διαρκώ ενημερό το Κοινοβούλιο για όλα τα στάδια τη διαδικασία. Στι περιπτώσει του Προέδρου τη Τραπεζική Αρχή, ε, λόγου χάρη, και του μέλου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νέου Μηχανισμού Εξυγένση, πολλοί υποψήφοι, μεταξύ των οποίων γυναίκε, δεν πέρασαν ε, τα διάφορα στάδια επιλογή. Δεν είχαν ελάχιστα, ε, απαιτούμενη ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία ή την ε, μακροχρόνια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών που απαιτεί το. Γι' αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε τι συνεννοήσει μα με το σώμα σα για το πολύ σημαντικό αυτό ε, θέμα. Στι περιπτώσει όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει στην όλη διαδικασία, θα συνεχίσουμε να τον διαδραματίζουμε και να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ισότητα των φύλων. Όταν θα συνθέτουμε τον κατάλογο υποψηφίων για τι αρχέ και του οργανισμού παρακολούθηση των χρηματικών και Οικονομικών Υποθέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιούραβα. Για 1,5 λεπτό το λόγο τώρα έχει η κυρία Ντελάνγκε. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Μου έχει κοπεί λίγο η ανάσα γιατί μόλις έφτασα έτρεχα. Λυπούμε που άκουσα τα μισά μόνο από αυτά που είπατε. είχα κάποια επικοινωνία. Ε, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, οι γυναίκες να μπορέσουν να τα συμφιλιώσουν όλα. Ε, να συμφιλιώσουν την οικογενειακή και την επαγγελματική τους ζωή. Σε ό,τι αφορά τους διορισμούς που είναι το θέμα μας, πραγματικά πρέπει να υπάρξει ε, ισορροπία Παραδείγματος χάρη ε, τι γίνεται ε, στην Ιταλική αντιπροσωπεία ε, όταν έχουμε να διορίσουμε κάποιον στη θέση του ESM για παράδειγμα στο μηχανισμό σταθερότητας και υπάρχει και μια Ιρλανδή γυναίκα η άλλη υποψήφοι είναι δύο πώς γίνεται η επιλογή είναι μια συμβολική συζήτηση ουσιαστικά αυτή που κάνουν θα πρέπει να λύσουμε πραγματικά το, το ζήτημα αυτό. Στα υψηλά αξιώματα ε, είναι λίγες οι γυναίκες που έχουν πραγματικά πάρα πολλά προσόντα που θέτουν υποψηφιότητα. Εκεί πρέπει να δράσουμε, στις τράπεζες, ε, στο επίπεδο των επιχειρήσεων, στο επίπεδο της πολιτικής, ε, να δώσουμε τη δυνατότητα σε περισσότερες γυναίκες να καταθέσουν υποψηφιότητα για θα τους έχουμε εξασφαλίσει ε, την με καλύτερη συμφιλίωση της επαγγελματική και οικογενειακής τους ζωής. Διότι αν μια γυναίκα έχει 6-7 χρονών παιδί, είναι δύσκολο ή παραδείγματος χάρη αν στο σχολείο ρωτήσει κανείς ε, πώς φαντάζεστε έναν πυροσβέστη ή έναν ε, χειρουργό, ε, φαντάζονται στο 60-70% ότι θα έρθει στην αίθουσα να τους κάνει παρουσίαση ένας άντρας, ένας αστροναύτης για παράδειγμα. Και εκπλήσονται βλέποντας να έρχεται μια γυναίκα. Δεν τις φαντάζονται τις γυναίκες αυτού του ρόλου. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπρέσο έχει τώρα το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα όπως εδώ σωστά υπενθυμίστηκε, η διαδικασία ε, επιτέλους ε, ορθώς ολοκληρώθηκε. Θα ψηφίσουμε, δεν είναι θέμα αυτό. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ πιο περίπλοκο. Όλος ιδιαίτερος και όπως θύμισε η Επιτροπός, έχουμε να κάνουμε με υπεκπροσώπηση των γυναικών σε όλα τα όργανα και τα υψηλα, τις θέσεις υψηλών στελεχών, σε όλα τα επίπεδα και στις ιδιωτικές όμως εταιρείες. Αλλά το ίδιο και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα χρηματοοικονομικά, ε, η υποεκπροσώπηση αυτή είναι ακόμα πιο έντονη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι πώς θα αντιστραφεί αυτή η τάση. Διότι αν υποψηφιότητες ε, δεν υπάρχουν, καταλαβαίνω δεν έχουμε και επιλογή. Όμω πολλέ φορέ υπάρχουν υποψήφια γυναίκε και δεν διευκολύνονται οι σταδιοδρομίε των γυναικών στα όργανα αυτά. Τι να πούμε δηλαδή στα κορίτσια να σπουδάζουν οικονομία για να μην ε, έχουν επαγγελματική σταδιοδρομία ε, αξιοπρεπή. Διότι όταν κάνουν σπουδέ οικονομολογία, τι να του πούμε, δεν θα πάτε μπροστά, θα πετύχετε ένα τίποτα. Τελικά έτσι δεν θα έχουμε αποψηφιότητε. Αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Άρα ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο να παρακολουθεί την ορθότητα των διαδικασιών, αλλά να προωθήσει και την ορθότητα ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη παρουσίαση των σπουδών σε θέματα τεχνικά, οικονομικά, επιστημονικά για τι γυναίκε, εάν θέλουμε να έχουμε υποψήφιε γυναίκε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Τρεμπέσιος, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε στο Βραδεμβούργο αποφασίσαμε ότι στο μέλλον ε, στο ε, Κοινοβούλιο ε, θα έχουμε μια, ένα μέτρο ώστε να δώσουμε βάση ε, στην ισότητα των δύο φύλων, όπως ε, έχουμε και στο εκλογικό σώμα 50% ε, άνδρες και 50% γυναίκες, θέλουμε το ίδιο να αντικαθρεπτίζεται και στο κοινοβούλιο, δηλαδή στην πολιτική να έχουμε το ίδιο επίπεδο συμμετοχής ανδρών και γυναικών, κάτι το οποίο υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, σε τρεις ε, ε, εκδηλώσεις που πήγα είδα ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο έδαφος που πρέπει να καλυφθεί. Θα πρέπει λοιπόν απ' την άλλη να δούμε πού σταματάει και το fair, το δίκαιο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη εκπροσώπηση, αλλά υπάρχουν και πολλές άλλες ε, μειονότητες. Υπάρχουν χριστιανοί, μουσουλμάνοι, υπάρχουν άνθρωποι με διαβήτη, υπάρχουν άνθρωποι με αναπηρία, υπάρχουν ομοφιλόφιλοι. Υπάρχουν, λοιπόν, υπάρχουν κάποια όρια κάπου πρέπει να μπουν ε, σε όλες αυτές τις ποσοστώσεις και σε όλες αυτές ε, τις ε, ισορροπίες. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τους πολίτες μας και να διαλέξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις καλύτερες δεξιότητες που ε, είναι ουσιαστικά ε, αυτοί που από πλευράς ποιότητας είναι πλέον κατάλληλοι. Ε, και εγώ ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια σε τεχνικές σπουδές. Τις σπουδές μου ήταν ένα 15% οι γυναίκες. Δεν έχει αλλάξει το ποσοστό αυτό, η αναλογία αυτή. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι γυναίκες είναι διαφορετικές από του άντρε. Τα δύο φίλων είναι διαφορετικά. Ο κύριο Τόρβαλ, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Στην τελευταία δήλωση Συμβουλίου Επιτροπής ακούσαμε τα τελευταία προσχήματα. Μας είπαν δηλαδή ξανά ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Περιγράφουμε και πάλι το πρόβλημα, λέμε ξανά ότι υπάρχουν γυναίκες με γνώση σε υψηλό επίπεδο και ότι αυτές προχωρούν. Ε, κι όμως, συγγνώμη, υπάρχει πρόβλημα. Παρά τις εξηγήσεις αυτές και τα προσχήματα. Λέει δηλαδή, κάθε φορά που καθυστερεί ένα αεροπλάνο, ναι, καθυστερεί γιατί καθυστέρησε επειδή καθυστέρησε, επειδή άρχισε να φτάσει στο αεροδρόμιο και αυτό είναι η αιτία της καθυστέρησης της αναχώρησης. Ευχαριστώ πολύ. Θέλουμε κάτι περισσότερο από αυτό. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η κυρία που μίλησε προηγουμένως, η συνάδελφος, είπε ότι ναι, υπάρχουν διαφορές στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο. Εγώ πάω πίσω στην κρίση του 2008, όταν όλες οι τράπεζες ήταν υπό τη διοίκηση ανδρών. Άνδρες αποφάσισαν την εποχή εκείνη. Αυτοί πήραν τις αποφάσεις. Αυτοί οδήγησαν στην κρίση. Χρειαζόμαστε λοιπόν σίγουρα περισσότερες γυναίκες επικεφαλής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Τόρολτ. Κύριο Γκίγκολτ έχει το λόγο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι προτάσει Κομισιών, και, Κομισιών και Συμβουλίου για την ισορροπία των φύλων κατά το Διερισμό σε ενωσιακές θέσεις του οικονομικού και νομισματικού τομέα. Ε, είναι, θα έλεγα, ε, αναχρονιστικές, με την έννοια ότι δεν ζούμε πλέον ε, στον 20ο αλλά στον 21ο. Δηλαδή δεν είναι πλέον <laughs> οι γυναίκες διαφορετικές από του άνδρες, όπως είπε μια προλαλή σα. Εδώ και καιρό έχουν αξιώματα ε, υψηλά ε, οι γυναίκες και στον τομέα των οικονομικών και των νομισματικών και πάρα πολύ δικαιολογημένα και σωστά. Και στα κοινοβούλια οι γυναίκες δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια ε, και γι' αυτό παρακαλώ να είμαστε και εμείς συνεπείς εδώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι θέμα ε, του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό το οποίο πρέπει να βρεθεί ε, από Συμβούλια και Κομισιό είναι να σταματήσει να ισχύει μια μεσαιωνική πρακτική για το διορισμό ε, σε ενωσιακές θέσεις, κάτι που δεν αντακατοτρίζει την πραγματικότητα. Κυρία Ματίας τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η ισότητα παραμένει δυστυχώς νεκρό γράμμα όταν ε, μιλάμε για τις θέσεις στον οικονομικό και νομισματικό τομέα. Πού είναι οι γυναίκες? Έχουμε διάφορες οδηγίες, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει ισχνό. Οι γυναίκες είναι ελάχιστες η Κομισιόν ούτω ή άλλω υποβάλλει ξανά του τελικούς καταλόγους υποψηφίων οι κυβερνήσει των ε, ευρωπαϊκών κρατών δεν έχουν γυναίκε άξιε με προσόντα που να έχουν απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη. Αυτό είναι προσβολή για τι γυναίκε. Είναι προσβολή για όλου. Ε, είναι μια προσβολή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι όνειδο. Πραγματικά ελπίζω ότι όταν κάποια στιγμή ξαναπαρουσιαστούν υποψήφοι για του οργανισμού σα και έχουν μόνο άντρε, αυτό το σώμα που υποτίθεται ότι υπερασπίζεται την ισότητα των φύλων θα του απορρίψει. Γιατί πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη και ισότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτέλου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ματίας. Δυόμιση λεπτά κυρία Ντορνανό. Πρόεδρε, την 3η 26 Φεβρουαρίου τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ είχαν ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Φίλιπ Λαν, προεπιλέγεντα ως μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, με τον κύριο Καμπά, Επικεφαλή τη ε, Τραπεζική αρχή και τον κύριο Σεμπαστιάν Λανό Λαβιόλα για τη θέση του μέλου του Συμβουλίου του Ταμείου Ξηγήρησης Τραπεζών. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Οι γυναίκε δεν εκπροσωπούνται παρκώς στι ανώτερες θέσει στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Και αυτό δεν με εκπλήσει. Όταν ξέρουμε ότι μόνο 39% των θέσεων, των διοικητικών θέσεων στα ευρωπαϊκά όργανα ανήκουν σε γυναίκες. Μας αρέσει το θέμα, συζητάμε και ξανασυζητάμε, αλλά όταν έρχεται η στιγμή να δράσουμε, να λάβουμε αποφάσεις, εξαφανιζόμαστε όλοι. Η ίδια η Κομισιόν στις Βρυξέλλες επί 13 προέδρων τα τελευταία χρόνια ούτε μία γυναίκα. Ούτε μία γυναίκα επίση, μεταξύ των ιδρυτικών πατέρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Επί 28 επιτρόπων μόνο 9 γυναίκε. Σα φαίνεται φυσικό αυτό? Από τα 250 εκατομμύρια γυναίκε τη Ευρωπαϊκή ένωση δεν βρέθηκαν 14 ικανέ γυναίκε, προφανώ και όχι. Όλα αυτά γίνονται επισκοπών. Και το λέω αυτό για να αποδείξω γιατί είναι έτσι τα πράγματα και στον οικονομικό τομέα. Δείτε τον κύριο Γιούνκερ. Η κυρία Περιά Σολίν είναι επικεφαλής της ε, εθιμοτυπίας και εγώ διαρωτώ με. Αυτό είναι το παράδειγμα που θέλουμε να δείξουμε. Αυτή είναι η εικόνα της γυναίκας για την Επιτροπή Γιουνκέρ. Οι φιλοευρωπαϊστές υπενθυμίζουν πάντοτε ότι μία από τις βασικές αρχές, μια αρχή του 57, είναι η ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών. Και όμω τόσα χρόνια μετά, οι ανισότητες στον τομέα των αμοιβών είναι εξόφθαλμες και μάλιστα ακόμη περισσότερο στις χώρες που είδησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιτέλους, ας λάβουμε συγκεκριμένη δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Αντορνανό. Το λόγο έχει ο κύριος Για ένα λεπτό. για μια ακόμη φορά γιορτάζουμε αυτή την αρρωστημένη ψύχωση ε, για την ισότητα και δείχνετε ότι έχετε ε, χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και ένα νήπιο ε, θα έχει μεγαλύτερη λογική από τους ευρωβουλευτές που αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες ε, σε θέσεις ψηλές και εσείς επιμένετε. Επιμένετε, γνωρίζετε δηλαδή καλύτερα και από τις ίδιες τις γυναίκες. Είναι γελίο το όραμα που έχετε για τις γυναίκες. Λέτε ότι είναι το μισό εκλογικό σώμα γυναίκες. Και λοιπόν... Υπάρχουν και ανήλικοι που δεν εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ακόμα. Και τι θα πει και αυτό λοιπόν. Ε, είναι και αυτοί άτομα που τη διακριτική μεταχείριση. Μήπως να δούμε τι γίνεται ε, με την ισορροπία των φίλων ας πούμε, στη θέση των οδηγών και των διερμηνέων. Έχουμε πολλές γυναίκες διερμηνές. Πώς πρέπει να τις πάμε να γίνουν σοφέρ. Υπάρχει, λέει ο Πρόεδρος, ε, μία ερώτηση, μία ε, μπλε κάρτα. από την κυρία Βάτμανς. Τη δέχεστε, κυρία Βάτμανς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι οι γυναίκες που είμαστε εδώ σήμερα στην αίθουσα έχουμε ε, αγανακτήσει με αυτά που ε, μόλις ακούσαμε. Είναι απίστευτα αυτά που βγήκαν από το στόμα σας ε, για το κοινοβούλιο, για τους βουλευτές που λέτε ότι δεν είμαστε έξυπνοι, δεν έχουμε ευφυΐα και δεν καταλαβαίνουμε. Θέλετε πραγματικά να εκπροσωπήσετε εδώ τις γυναίκες. Ερώτηση έπρεπε να κάνετε, κυρία Βάουταν. Και μέχρι τα 27 δευτερόλεπτα δεν είχατε κάνει ερώτηση. Δεν έχω ελπίδα ότι θα κάνετε ερώτηση. 30 ε, δευτερόλεπτα ε, ουσιαστικά ε, διαρκεί η παρέμβαση στο πλαίσιο της μπλε κάρτας, αλλά μόνο για ερώτηση δίνουμε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε την ερώτηση σας πάρα πολύ σύντομα. Με μικρόφωνο, παρακαλώ. Εντάξει. Θα θέλατε παρακαλώ να επαναλάβετε τη δήλωσή σας ότι πιστεύετε ότι είναι λιγότερο κατάλληλες ε, οι γυναίκες γιατί αυτά κατάλαβα να ε, για υψηλά αξιώματα δηλαδή από αυτά που είπατε. απάντηση. Εγώ είπα ότι ε, λογική δεν έχουμε, κοινό νου. Δεν είπα ότι δεν ε, είναι έξυπνοι βουλευτέ και φυσικά οι γυναίκε είναι πιο κατάλληλε για κάποιε θέσει, για κάποιε δουλειέ και οι άνδρες πιο κατάλληλοι για άλλε δουλειέ. Οι διερμηνεί παραδείγματο χάρη, σε μεγάλο βαθμό είναι γυναίκε, άρα μάλλον είναι πιο κατάλληλε οι γυναίκε για τη δερμηνία και υπάρχουν πολύ περισσότεροι οδηγοί, σοφέρ, άρα μάλλον είναι καλύτεροι σε αυτό από τι γυναίκε. Πρέπει να το δεχτούμε. Τα ταλέντα διαφέρουν. Ευχαριστώ. Ε, Επέτρεψα μία ε, μπλε κάρτα και είμαι και λιγότερο αυστηρός, θα έχετε παρατηρήσει μέχρι στιγμής ό,τι αφορά ε, το χρόνο αγόρευσης. αλλά δεν ήμουνα γενναιόδωρος απέναντι ε, στην κυρία Ντελάγκεν. Ο κύριος Φέρμπερ για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι το ότι δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των δύο φύλων σε ό,τι αφορά την Κεντρική Τράπεζα ή τα άλλα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μυστικό ε, και αυτό ε, βασίζεται και στο τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο, ότι και εκεί δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Ε, Επομένω, είναι δύσκολο να υπάρξουν διαθέσιμε γυναίκε για υψηλά ενωσιακά αξιώματα. Άρα και σε εθνικό επίπεδο, στι εθνικέ δομέ θα πρέπει να βρουν θέση οι περισσότερε γυναίκε. Και αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Αυτό το οποίο με ενοχλεί όμω εδώ είναι η υποκρισία με την οποία γίνεται αυτή η συζήτηση. Έχουμε ε, κάποιε πολιτικέ ομάδε που εξεγείρονται και εξανίστανται. Είχαν όμω τη δυνατότητα σε ό,τι αφορά τον Ευρωπαϊκό Επιτροπτικό Μηχανισμό. Θα είχαν τη δυνατότητα να, να εκλέξουν μια γυναίκα και αυτοί λοιπόν που ε, εδώ πέρα διαρριγνούν τα ημάτια του ε, ε, διάλεξαν έναν άντρα. Ε, λοιπόν, τι μιλάμε τώρα για την ε, ε, ισότητα των δύο φύλων. Στείλανε email και γράφανε ε, διάφορα. Ε, πραγματικά δεν έχω ξαναδεί ε, τέτοια διακριτική μεταχείριση ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό παρακαλώ τους συναδέλφους όταν έχουμε τη δυνατότητα να εκλέξουμε, να διορίσουμε μια γυναίκα να το κάνουμε και όχι να έχουμε εδώ αυτή την υποκριτική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να λέμε έμπτα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γετεμάκη, για ποιον ε, είναι η μπλε κάρτα. Για τον κύριο Σόσνερ ή για τον κύριο Φέρμπερ. The... Παναλαμβάνω, για ποια παρέμβαση θέλετε για τον κύριο Σόσνερ. Δεν μπορώ να δεχτώ την μπλε κάρτα για προηγούμενο μιλητή. Κυρία Μπερέση, τώρα το για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο περίπου, στις 8 Μαρτίου πέρσι, ο πρόεδρος του σώματος έγραφε στα ευρωπαϊκά θεσμικά οργανά του επικεφαλής του μετά τον διορισμό του κυρίου Δεκίτος ε, και μετά την, ε, το διορισμό στην Κεντρική Τράπεζα έλεγε ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλογο υποψηφίων με τρία ονόματα τουλάχιστον και ισορροπία των φίλων. Δεν έγινε αυτή τη στιγμή καν κάτι τέτοιο όταν προτάθηκε ο κύριος Φίλιπ Λέιν και ε, περιμένουμε να δούμε τι θα κάναν το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και, το, και η Επιτροπή για την προσπάθειά του αυτή για του μελλοντικού διορισμού. Σε σχέση με την επιστολή αυτή, μα λέτε όλοι ότι ο ρόλο σα είναι περιορισμένο, αλλά μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση. Διότι κάποια στιγμή η κατάσταση αυτή γίνεται απαράδεκτη. Και η στιγμή αυτή έχει φτάσει. Δεν είναι φυσιολογικό στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στις, ε, ε, στις, ε, στους φορείς που ασχολούνται με τα οικονομικά θέματα, να μην γίνεται καμία προσπάθεια να γίνει σε αυτό γίνει σεβαστή ισορροπία των φίλων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Πρέπει να αλλάξετε λοιπόν το πλαίσιο, ε, την οτροπία. Στο επόμενο κοινοβούλιο, στην επόμενη θητεία, κάθε μέλο θα πρέπει για τη θέση επιτρόπου να προτείνει τουλάχιστον έναν άντρα υποψήφιο και μια γυναίκα υποψήφια για να υπάρχει έστω ισότητα στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ίδιο στι θέσει ευθύνη στα ε, στους, στους ε, οικονομικούς μας οργανισμούς θα πρέπει να υπάρχει κατάλογο υποψηφίων με ισορροπία των φύλων. Θα πρέπει επιτέλους να φτάσει η ώρα που το Κοινοβούλιο θα αναλάβει τις ευθύνες του για το θέμα αυτό. Ακούω το ΕΛΚ να δίνει μια ιδιαίτερη μάχη για να ε, πηρύψει ευθύνε στους σοσιαλιστέ και δημοκράτες για το θέμα αυτό. Γιατί και καλά η επιλογή ε, δεν ε, έγινε την κρίσιμη στιγμή και να προωθηθεί μια γυναίκα στην κατάλληλη θέση. Μα δεν νομίζω ότι η λογική θα πρέπει να είναι ότι εκ των προτέρων θα πρέπει να έχουμε επιλέξει γυναίκα. Δεν θα πρέπει να κατηγορείται η δική μα ομάδα για την κακή αυτή επιλογή. Όμως Ε, επειδή το θέμα των διορισμών θα συζητηθεί και την επόμενη Πέμπτη, θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά για τι διαδικασίε που θα επικρατούν στους οικονομικού οργανισμού. Συγγνώμη ε, που ε, δεν αφήνω παραπάνω να μιλήσετε. Ο κύριος Πιωτρόφσκι από το ECR το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, συναδελφοί. Σήμερα μιλάμε για την ισότητα ενώψη τριών διορισμών στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων. Εμείς θα κληθούμε να εγκρίνουμε τους διορισμούς του τελικού καταλόγου. Εμείς ως ECR είμαστε υπέρ της ισότητας των φύλων, όμως θέλουμε και μια γεωγραφική ισορροπία. Όλοι οι υποψήφοι είναι προκειμένο από τις χώρες της λεγόμενης παλιάς Ευρώπης. Πού είναι η Ανατολική Ευρώπη? Και δεν νομίζω να υποστηρίζει κανείς ότι δεν έχουμε κανούς υποψηφίους. Ας μην ξεχνούμε, επίσης, ότι όλοι οι υποψήφοι πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα. Φαντάζομαι αυτό ισχύει. Το φύλλο λοιπόν δεν είναι ούτως ή άλλως η μόνη παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη. Να προσθέσω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή έχει 28 επιτρόπους, 19 γυναίκες και μόνο 9, 19 με συγχωρείτε άνδρες και 9 γυναίκες. Και αυτό είναι ένα σημάδι, είναι μια ένδειξη ότι δεν ισχύει πλήρως τουλάχιστον το δικαίωμα της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όμως το θέμα είναι αυτό. Όταν μιλάει λοιπόν η Κομισιόν, α κοιτάξει πρώτα τον εαυτό της. Ευχαριστούμε κύριε Πιοτρόφσκι. Ένα λεπτό, η κυρία Ιντφέλντ. Yes, um, thank you, chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σόσνια, απέδειξε πέραν πάση αμφιβολίες γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε την ευθύνη του κόσμου στου άνδρε. Το έχουμε συζητήσει τόσες φορές και κάθε φορά ακούμε τα ίδια επιχειρήματα. Κάποιοι λένε ας προχωρήσουμε έτσι όπως είναι τα πράγματα, αλλά την επόμενη φορά, πραγματικά την επόμενη φορά θα έχουμε μια ισόρροπη λύση με άνδρες και γυναίκες σε ίσους αριθμού. Ε, αυτά τα πράγματα δεν πιστεύουμε πια. Το θέμα δεν είναι ποιοι είναι καλύτεροι, αν άνδρες καλύτεροι, οι γυναίκες καλύτερες. Το θέμα είναι ότι ποικιλία. Οι μεικτές ομάδες αποδίδουν καλύτερα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Και εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Την διακυβέρνηση των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων. Εδώ θα πρέπει να επιδιώξουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα. Ομάδα όμω, μια πραγματική ομάδα. Και κάποιοι θα πούν για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε αρκετέ ε, γυναίκε υποψηφίου, ικανές υποψηφίους Είμαστε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση 500 εκατομμυρίων ανθρώπων και μας λέτε ότι δεν υπάρχουν τρεις γυναίκες. Ε, τελευταία πρόταση, Πρόεδρε. Και δεν υπάρχουν τρεις γυναίκες ικανές στο επίπεδο αυτό. Ε, ευχαριστώ. Διακόπτε ο Πρόεδρος. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό λέγω. Έχει το... Κύριε Ιντφέλτ και κύριε Φέρμπερ, ενδιαφέρουσα η ενθερμό αυτή ανταλλαγή απόψεων, αλλά δεν ε, ακουγόταν ε, γιατί τη διερμηνία, άρα πέρασε έτσι. κυρία Σκοτ Κέιτο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Τι σημασία έχει ε, που υπερτερούν οι άντρες στον οικονομικό τομέα. Μήπως γιατί έχουν τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, σχεδόν το μισό ε, περιουσιακά στοιχεία, 8, ε, στα χέρια 8 ανδρών. Ε, οι άνδρες κάποιες φορές παραγνωρίζουν το ρόλο της γυναίκας, της μητέρας, των δασκάλων κτλ. Το θέμα είναι όχι αν είμαστε καλύτερες χειρότερες. Απλά πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι οι, μισές, οι μισοί άνθρωποι του πλανήτη που είναι γυναίκες πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και αυτό να αντικατοπτρίζει και στα υψηλά αξιώματα. Εγώ δεν θα ε, συνεχίσω να συμμετέχω ε, σε αυτή την υποκριτική παράσταση, μόνο λόγια και όχι έργα. Σε ό,τι αφορά ε, τους ευρωπαϊκούς αποπτικούς οργανισμούς, τουλάχιστον στον κατάλογο προεπιλογής να περιλαμβάνεται μια γυναίκα. αλλιώ, δεν θα ξανά ε, ψηφίσουμε εμείς. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, Βιέγας. Ευχαριστώ. Το θέμα αυτό εγείρει δύο προβληματισμούς. Πρώτα απ' όλα, την ισότητα των φίλων, που εμφανώς δεν ε, γίνεται σεβαστή στις αρχές εποπτείας ή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως, έχει και ένα άλλο ζήτημα το θέμα της δημοκρατικής ε, λογοδοσίας και παρακολούθησης της λειτουργίας αυτών των οργανισμών. Ε, για παράδειγμα, όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήταν ένα όργανο ε, πολιτικός ουδέτερο, με τεχνικέ αρμοδιότητε. Όμω, με το πέρασμα των χρόνων, είδαμε τι διαστάσει πήρε στο, στο, στα πλαίσια του προγράμματο λειτουργία τη Κεντρική Τράπεζα. Δεν προβλέφθηκε όμω καμία δημοκρατική λογοδοσία. Αν θέλουμε να είμαστε λοιπόν σοβαροί, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην επιλογή των υποψηφίων, των ε, διοικητικών στελεχών των θεσμών αυτών, δεν μπορεί να περνά από μια κλειστή διαδικασία, από, ε, ένα, ε, από διαδικασίε και κλεισμένων των θυρών. Οι κατάλογοι των υποψηφίων πρέπει να παρουσιάζονται και να έχουν ε, τουλάχιστον κάποιο όνομα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει καμία παρουσία γυναίκας. Τη στιγμή που ήρθε στα χέρια μας ο κατάλογος των υποψηφίων, ε, τελικά δεν ε, έλαβε υπόψη της καν την τελική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου. Η τελική παρουσίαση κάποιων ε, διαδικασιών λοιπόν στα θεσμικά όργανα είναι ακατανόητη, είναι αντιδημοκρατική και είναι τελείως αδιαφανής η λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ε, ουσιαστικά κινούνται από τα χρήματα οικονομικά συμφέροντα και δεν υπάρχει κανένα, καμία διάσταση δημοκρατικής παρακολούθησης. Ευχαριστούμε κύριε Βιαγάς. Με 1,5 λεπτό. Κυρία Εστάρα Σφεραγκούτ. Ευχαριστώ. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γυναίκα, μία γυναίκα μάλλον στην Εκταλιστική Επιτροπή μεταξύ πέντε ανδρών. Στο Γενικό ε, στο Συμβούλιο πάλι μία μεταξύ Στι εποπτικές αρχές. Άνδρες όλοι οι πρόεδροι. Ε, και στην αρχή εξυγίανση των τραπεζών. Πάντα, πάλι μόνο άντρε. Στον εποπτικό μηχανισμό, πρόεδρο άντρα. Τρει ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ πρόεδρος άντρα. Ε, άρα είναι σαφές ε, ότι υπάρχει ανισότητα ε, στις θέσεις ισχύω. και το βλέπουμε αυτό και στις υψηλές θέσεις στον οικονομικό, χρηματοπιστωτικό, νομισματικό τομέα. Όμως μια από τις αρχές ένωσης είναι η ισότητα των δύο φύλων. Πρέπει να είναι οριζόντια και εγκάρση η αρχή της ισότητας. Η ισότητα σημαίνει περισσότερη δημοκρατία, σημαίνει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει μια ρήξη να καταρριφθούν τα στερεότυπα που ανέφερε και ο κύριο Σόσνιερ τελικά ε, και θα πρέπει να ε, εκπαιδεύσουμε μια κοινωνία ισότιμη δίκαιη ε, που θα στην πράξη θα εφαρμόσει την ισότητα των δύο φύλων. Ευχαριστούμε πολύ. Επιτρέπετε ερώτηση από τον κύριο Σόσνιερ, κυρία Σταράς. Δέχεστε. Ναι. Κύριε Σόσνιερ. Ε, ε, ε, Με συγχωρείτε, αλλά θα δείτε στατιστικές αν κοιτάξετε στο YouTube ποιος παρακολουθεί τι. Έχει ποσοστά. Τα πολιτικά φιλμ κατά 80% τα κοιτάζουν άντρες. Και αυτό δεν είναι γιατί ο κακό και δαιμονικό Όσνιερτ αποφάσισε να απαγορεύσει στι γυναίκε να κοιτάζουν αυτά τα φιλμ. Οι γυναίκε δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Δεν ήταν ερώτηση αυτό, κύριε Σόσνη. Było pytanie, zapytałem, co pani zamierza zrobić z tym, że kobiety nie oglądają filmów na o tematyce politycznej. Όχι, εγώ ρώτησα, τι θα κάνετε για το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν βλέπουν πολιτικά φιλμ στο YouTube, ας πούμε, πώς θα τις υποχρεώσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ντροπή και όνειδος που ε, είστε, έχετε μια έδρα ε, στον οίκο της ε, ειρήνης και των ευρωπαϊκών αξιών. Εσείς. Είναι ντροπή. Ευχαριστώ κύριε Στάρα Αργκούτη. Για ένα λεπτό κυρία Τόγια. Δεν θέλω να χάσω ούτε ένα δευτερόλεπτο από το λεπτό μου, αλλά πρέπει να το κάνω για να εκφράσω τον αποτροπιασμό μου και το όνειδο που αισθάνομαι με τέτοια λόγια ντροπή που ακούγονται από το Κοινοβούλιο όταν εκφραζόμαστε για το θέμα των γυναικών. Πραγματικά είναι σαν να έχουμε ετηθεί. Θα πρέπει επιτέλου ε, την ε, θητεία μα να την ε, οδηγήσουμε και σε ένα αίσιο πέρα. Προσπαθούμε να κάνουμε να ακουστεί η φωνή μα και δεν μα ακούει. Η Επιτροπή λέει ότι μα ακούει, δεν ακούει το Συμβούλιο και τούμπαλιν. Θα πρέπει λοιπόν κάτι να γίνει με τι γυναίκε. Δεν είναι αφηρημένη η έννοια τη ισότητα. Θα πρέπει να την προασπιστούμε πιο ε, πραγματικά, γιατί μερικέ φορέ τα θεμέλια των αξιών είναι λίγο θεωρητικά και φιλοσοφικά. Είναι θέμα γενικού συμφέροντο, είναι πρακτικό. Θα πρέπει να μην το δούμε ω μια πράξη καλή θέληση ή δεν είναι μια χειρονομία ευγένεια. Είναι θέμα ε, που έχει να κάνει με το ότι η παρουσία των γυναικών στου θεσμού ε, ενισχύει, κάνει πιο πιο εύρωστο στους θεσμούς. Να αναφέρω μια μελέτη από την κόρτ τον ε, Οργανισμό Ελέγχου των Κρατικών Φορέων τη Ιταλία. Δείχνει επιστημονικά ότι οι κοινωνίες που ε, η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια είναι μεγαλύτερη μπορούν να αντισταθούν καλύτερα στις περιπτώσεις κρίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τόγια. Κύριε Σουρτασούν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταδικάζω περίφραστα τα λόγια ε, που ακούσαμε ότι δεν μπορούν οι γυναίκες να είναι ε, οδηγοί, οι άντρες να είναι διερμηνείς. Δεν υπάρχει πιο φαλοκρατικό σχόλιο. Πραγματικά ντρέπομαι. Το θέμα αυτό ε, που μας απασχολεί δεν μπορεί να έχουμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στα εποπτικές αρχές, μόνο άνδρες. Και ήταν δύο γυναίκες οι οποίες είχαν αξιώσει που φεύγουν και θα αντικατασταθούν και αυτές από άνδρες. Ε, και πραγματικά έχουμε ζητήσει να έχουμε ε, καταλόγους ε, όπου εκπροσωπούνται ισότιμα τα δύο φύλλα για να κάνουμε την επιλογή. Και αυτό δεν γίνεται. Έπειτα έχουμε κινητοποίηση μαζική των γυναικών και την επέτειο, μάλλον την ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου. Πραγματικά αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς αυτή τη βδομάδα να μπλοκάρουμε αυτούς τους ορισμούς και να ζητήσουμε να μας στείλουν άλλη πρόταση. Ευχαριστούμε κύριε Σόσνιερ λέει ο πρόεδρος. Όχι, ευχαριστώ κύριε Ούρτασούν, κύριε Σόσνιερ Δεν θα σας επιτρέψω ε, την μπλε κάρτα. Ε, κύριε κυρία είναι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Μιλούμε για διορισμούς γυναικών σε υψηλέ θέσει. Όπω είπε και προλαλή σα, ναι, μα λένε την επόμενη φορά θα τα βρούμε. Μετά μας λένε, μα πώς θα βρούμε ικανές γυναίκες στον τομέα αυτών, είτε τον δημόσιο, είτε τον ιδιωτικό, στον οικονομικό και νομισματικό τομέα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής δεν υπάρχει δυνατότητα ισότητα. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει δυνατότητα ισότητα στο επίπεδο αυτό. Το θέμα βεβαίω είναι η ποιότητα των υποψηφίων. Θα παραγνωρίσουμε τις ικανότητες του μισού πληθυσμού της γης. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και θυμίζω τι γίνεται όσον αφορά την Επιτροπή. Πρέπει να υπάρχουν επίτροποι και επίτροποι, γυναίκε και άνδρε σε ίσου αριθμού. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε κυρία Πιετικάινεν. Για ένα λεπτό κυρία Πλίνκεβιτσιούτε. Ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, την Πέμπτη θα κληθούμε να ψηφίσουμε, να αποδεχθούμε, να εγκρίνουμε, να απορρίψουμε τους διορισμούς στα ανώτερα αυτά όργανα του οικονομικού και νομισματικού τομέα. Όλοι οι υποψήφοι προκειμένου είναι άνδρες. Οι γυναίκες δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Τόσο απλά. Μόνο 15% ήταν υποψήφοι. Ε, δεν μπορώ να αποδεχθώ ότι στον 21ο αιώνα πρέπει ακόμη να δίνουμε μάχη εμεί, οι γυναίκες για τις θέσεις αυτές. Όλα τα άλλα αποτελούν απλή παράβαση των βασικών μα αρχών και στον τομέα βεβαιω των ε, διορισμών προκειμένου. Η ισότητα είναι κατοχυρωμένη, όχι μόνο στις συνθήκες, αλλά και σε τρεις διαφορετικούς κανονισμούς που διέπουν και τη λειτουργία των εν λόγω οργάνων. Πώς είναι δυνατόν να παραβιάζει κατάφορα η Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια της την νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί να γίνει σεβαστή η αρχή αυτή της ισότητας και στον τομέα Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πλινκεβίτσι. Ούτε περνάμε στη διαδικασία προσέλκυσης προσοχής Προέδρου Φαρία, ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάνω απ' όλα για τα λόγια του κυρίου Σόσνερτ. Πρέπει να πω ότι θα πρέπει να απαγορεύονται τέτοιες εκφράσεις στο σώμα μας. Κυρία Επίτροπε, το Κοινοβούλιο μόνο να εκφράσει την δυσαρέσκεια του μπορεί για την διορισμό τριών ανδρών στα τρία υψηλά αξιώματα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα και των υπόλοιπων ε, θεσμών. Θα πρέπει να σεβόμαστε και την ισότητα των φίλων και τα ανθρωπινά δικαιώματα. Έφτασε η ώρα τι αρχέ και τι αξίε μα να τι θέσουμε σε εφαρμογή. Δεν μπορεί να επικρατεί αυτή η φαλοκρατική νοοτροπία υπέρ των ανδρών. Δεν αρκεί ότι οι άντρε αυτοί είχαν τα περισσότερα προσόντα. Τελικά δεν μπορούν πάντοτε αυτοί που έχουν τα περισσότερα προσόντα να είναι άντρε και σε αυτό το σώμα και σε άλλα ευρωπαϊκά όργανα και θεσμού. Θα πρέπει να επιλέγονται και γυναίκε για τι υψηλέ θέσει, τι θέσει ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δώσουμε ευκαιρίε για την ισότητα των φύλων και ε, στα οικονομικά ζητήματα και γενικότερα. Θα πρέπει να σκεφτείτε σε όλε τι υποθέσει πώ θα προωθείτε περισσότερο τι γυναικέ υποψηφιότητε και εσεί και στα κρατη Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κύριε Γκραπίνη. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε την ισορροπία των φύλων. Προφανώς η αρχή δεν είναι σύνθημα, είναι αναγκαιότητα. Και στον τομέα των οικονομικών και νομισματικών υποθέσεων. Εδώ η ευθύνη είναι κοινή. Λοιπόν, δείτε τι γίνεται στην Επιτροπή. Μόνο εννέα γυναίκες δείτε τι γίνεται στην ηγεσία των κρατών μελών. Λοιπόν, είναι θέμα παιδείας εν τέλει. Δυστυχώ έχουμε ακόμη άνδρες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άνδρες που δεν έχουν ενστερνιστεί τη βασική αυτή αρχή. Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Επιτροπή λοιπόν πρέπει να επιδείξουν διαφάνεια πρώτα απ' όλα και να αποδείξουν ότι οι προθέσεις τους είναι γνήσιες. δεν θέλουν να αρκεστούμε μόνο στους αντιπροέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μα ενδιαφέρουν και άλλες θέσει ευθύνη. Και εκεί πρέπει να ισχύσει η αρχή της ισότητας. Πόσε γυναίκες είναι ή υποδιοικητέ εθνικών κεντρικών τραπεζών. Α υλοποιήσουμε επίση αυτή τη γενική αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκραπίνη. Η κυρία Μπιλμπά Μπαραντίκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Αυτό το οποίο συνέβη με τους διορισμούς αυτούς ε, ε, σε οικονομικές θέσεις δείχνει ότι τελικά δεν ακούμε ε, τις ιαχές του 8 Μαρτίου τη αντιδράσεις των γυναικών που γίνονται όλο και πιο έντονες και όταν γιορτάσαμε το ευρώ, μόνο άντρε μίλησαν. Ελπίζω να μην συμβεί το ίδιο στα επόμενα 20 χρόνια. Εμεί θέλουμε μια πιο δίκαιη, πιο ε, δημοκρατική Ευρώπη. Θέλουμε ε, ταλέντο και χάνουμε εξαιρετικές υποψηφίους. Ε, πρέπει να σκεφτούμε σε αυτές, ε, αυτές τις γυναίκες και να τις προτείνουμε. Ε, θα είναι κάτι και αλλά είναι και υποχρεωτικό θα έλεγα. 8 Μαρτίου έλαβα στο τηλέφωνό μου μια εικόνα που τα έλεγε όλα. Ε, λένε ότι η επαγγελματική σταδιοδρομία είναι ένα στίβος. Δεν υπάρχουν εμπόδια ε, στο δρόμο των ανδρών, ενώ στο δρόμο των γυναικών είναι το πλυντή κτίριο, το ε, ψυγείο, ο φούρνος, ε, τα, ε, το σχολείο των παιδιών και λοιπά. Αυτό είναι το πρώτο που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, και νόμοι και αυτοκριτική. Διακόπτεται η κυρία Μπαραντίκ. Έθεριτς. Um, Ευχαριστώ. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι γυναίκες είναι τουλάχιστον εξίσου ικανές. Όμως, νομίζω ότι δεν χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη. Αυτοί που λένε ότι θέλουμε περισσότερες γυναίκες, να προσπαθούν να τις στηρίξουν με τρόπο τεχνητό. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι αν δουν περισσότερες γυναίκες στις θέσεις αυτές, θα το θεωρήσουν αυτομάτως πρόοδο στην προσπάθεια απελευθέρωση των γυναικών. Ε, και τώρα μήπως θα αρχίσουμε να ψάχνουμε τους άντρες τις θέσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι λύση. Έχουμε πολλές γυναίκες, ικανές γυναίκες, μορφωμένες γυναίκες, οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν ανώτερες θέσεις χωρίς να χρειάζονται σπρόξιμο ε, ούτως πίν για να φτάσουν στις θέσεις αυτές. Δεν χρειαζόμαστε αυτή την τεχνητή υποστήριξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Φέριτς, κυρία Γιατομάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Πίτη Κάινεν έκανε μια εξαιρετική παρέμβαση εδώ. Δεν είναι θέμα το να μην έχουμε αρκετές γυναίκες με προσόντα για τις θέσεις ευθύνη και τα υψηλά κλιμάκια της Κεντρική Τράπεζα και των άλλων θέσεων σε οικονομικού θεσμού. Το θέμα είναι ότι κάποιοι δεν θέλουν να δουν τι γυναίκε να προκόβουν. Λένε ότι δεν υπάρχουν αρκετέ γυναίκε με τα κατάλληλα προσόντα για τι θέσει αυτέ. Όχι. Πώ τολμάει να το λέει αυτό κανεί. Τι είναι αυτά που λέει ο κύριο Σόσνερτ. Είναι φρεχτά αυτά που ακούγονται εδώ πέρα για τι γυναίκε. Και κατά τα άλλα, είναι πολύ καλό να ακούμε εδώ διαφορετικές απόψεις, διότι κουβέντες σαν αυτές που ξεστόμησε ο κύριος Όσνιρτς είναι πια αρκετά κοινότοπες στην Ευρώπη. Εάν δεν υπήρχαν αρκετοί Σόσνιρτ, θα υπήρχαν και αρκετέ γυναίκε στι κατάλληλε θέσει. Αυτό έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιατεμάκη. Εδώ έκλεισε η διαδικασία προσέλκυση της προσοχής του Πρόεδρου. Παρά το ότι δεν το συνηθίζω, ε, θα πω κάτι. Ε, παρακολούθησα ε, πάρα πολύ προσεκτικά τη συζήτηση και τα προσυπογράφω όλα αυτά και πρέπει να πω ότι είναι μια συζήτηση που σπάνια φτάνει σε τέτοιες εκφράσεις και Στην, ε, στα αγγλικά υπάρχει μια πολύ όμορφη έκφραση chairman και chairwoman που δεν υπάρχει σε άλλες γλώσσες ε, και ε, τώρα μιλάμε όμως στο τρίτο ως chairperson ή ως chair. Έχουμε βγάλει ε, το ανθρώπινο στοιχείο από τον πρόεδρο ή την πρόεδρο ε, και αντί να, λέμε για, να μιλάμε ως chairman, chairwoman κτλ. μιλάμε ε, για την καρέκλα, chair. Κάναμε τον άνθρωπο αντικείμενο. Τέλος πάντων, η κυρία Γιούροβα έχει τώρα το λόγο. δεν ξέρω αν θα είναι λάθος, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω κάποια σχόλια Έχουμε αρκετές πολύ προσοντούχες γυναίκες στον οικονομικό νομισματικό τομέα. Όταν μιλάμε για αυτό το έλλειμμα πάντως, το βλέπουμε σε ό,τι αφορά τον τομέα της τεχνολογίας και πληροφορικής. Στον χρηματοπιστωτικό τομέα νομίζω ότι έχουμε αρκετές γυναίκες με ψηλά προσόντα. Το 62% των αποφύτων πανεπιστημίου που είναι γυναίκες